Αγαπητοί συναδελφοί, να περάσουμε στο τμήμα της συνεδρίασης της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων. Ευχαριστούμε τους, τους συναδέλφους από την Επιτροπή Απασχόλησης. Καλώς ορίζουμε εκ νέου τους προσκεκλημένους μας και εγκρίνουμε και την ε, ατζέντα της Επιτροπής Απασχόλησης τη Επιτροπή Οίκων, συγγνώμη. Θα επικεντρωθούμε λοιπόν τώρα στην άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα σχέδια δημοσιονομικών σχεδίων για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα σχέδια προπολογισμού. Δεν εντοπίστηκε κάποια σοβαρή περίπτωση μη συμμόρφωση. σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει κίνδυνο ε, μη συμμόρφωση. σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει και έχουμε και σε κάποια κρατημέλη ακόμα καθεστώς εντύπη, να σημειώσουμε ότι η Επιτροπή σύμφωνα και με τις συστάσεις αναχώρα, εξέφρασε πρόθεση να ασκήσει την διακριτική της ευχέρεια της οποίας ε, δικαιούται σύμφωνα με την οθομή ε, της νομοθεσίας για τις αξιολογήσεις. που αιτιολογούνται από τους δημοσιονομικούς στόχους για τη θεματική εφαρμογή του πίνακα από πλευρά μεθοδολογία θεωρώ ότι πρόκειται για μια θετική καινοτομία. για μια πιο εγκάρσια αξιολόγηση από πλευρά της Επιτροπής ε, του συνολική ε, οικονομική ε, στάση και των μακροοικονομικών όρων για μια πιο αντρή αξιολόγηση των συνθήκων. Συνολικά, ξέρουμε ότι υπάρξει σημειωτική μείωση και στο έλλειμμα και στη χρέωση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το έλλειμμα. Είμαστε φυσικά ακόμα πάνω από τους όρους μας, από τους στόχους μας. Αλλά οι προβλέψεις για το επόμενο επίπεδο χρέωσης είναι καλύτερες από την προηγούμενη. Έχουμε ακόμα δηλαδή μια μεγαλύτερη απόδοση από ό,τι περιμέναμε. Και υπάρχει και ιδιαιτερότητα σε ό,τι αφορά την δημοσιονομική στάση. Θετικά στοιχεία. Να δώσω λοιπόν το λόγο πρώτα στον Αντιπρόεδρο Ντομπρόψκης και στη συνέχεια στον κύριο Μοσκοβισή. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Αξιότιμοι βουλευτέ. Πέρα από το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και το πακέτο αυτού, εγκρίναμε γνωμοδοτήσει για τα σχέδια προϋπολογισμού για 28 κράτη-μέλη, για όλα δηλαδή, εκτός από την Ελλάδα που είναι ακόμα σε ε, το πρόγραμμα. Σε ό,τι αφορά και το Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη, οι γνωμοδοτήσει λοιπόν για τα σχέδια προπολογισμού αποτελούν μια σημαντική άσκηση για την επιτήρηση των ε, κρατών της Ευρωζώνης που επιτρέπει στα κοινοβούλια και στα εθνικά κοινοβούλια να λάβουν υπόψη τέτοιε συστάσεις κατά την έγκριση του οριστικού προϋπολογισμού. Στην Ευρωζώνη λοιπόν έχουμε αύξηση της ανάκαμψης και αναμένουμε να συνεχιστεί αυτή η ανωδική τάση. Ωστόσο, δεδομένου το ότι τα κράτη-μέλη βρίσκονται σε διάφορες φάσεις του οικονομικού κύκλου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει την ανάγκη να υπάρξει σωστή ισορροπία μεταξύ ε, υγεία των δημοσιονομικών και υποστήριξη ε, τη οικονομική ανάπτυξη, η μείωση τη υψηλή χρέωση και η δημιουργία αποθεματικών, δημοσιονομικών αποθεματικών είναι σημαντικό για να υπάρχει περιθώριο λιγμού σε περίπτωση επενδυτικών κρατασμών. Σε ό,τι αφορά τώρα των, τις μεταρρυθμίσει μεταρρυθμίσεις. Ε, μετά από μια ε, βελτίωση το 2017, η το διασφαλτικό έλλειμμα το 2018 αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,8% ποσοστό του ΑΕΠ. Η νομοσυνομική στάση της Ευρωζώνης είναι ευρέω ουδέτερο. Αυτό είναι το ευκταίο δεδομένου ότι η οικονομική ανάκτηση χαρακτηρίζονται από τέτοιες μελλοντικέ τάσει και αυτή η δεύτερη δημοσιονομική στάση συνάδει και με τις στάσεις του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Σώματος. Έχουμε μόνο δύο κράτη της Ευρωζώνης, την Ισπανία και τη Γαλλία, στη διαδικασία ε, υπερβολικού ελλείμματος που θα πρέπει να μειώσουν κατά από 3% του ΑΕΠ το ελλείμμα η Ισπανία και το σχέδιο προπολογισμού θεωρείται ότι συνάδει με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης σε γενικές γραμμές και προβλέπουμε το 2018 να είναι το έλλειμμα κατά από 3%, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε πετύχει αυτό το στόχο. Η Γαλλία υπερβολικό έλλειμμα φέτος και ως εκ τούτου θα μπει στο προληπτικό σκέλος ε, του Μηχανισμού Σταθερότητας και Ανάπτυξης από το 2018 και αν επαληθευτεί το σενάριο αυτό Τρέχει κίνδυνο να μην συνάδει με το GDP. Λίγα είναι τα κράτη-μέλη τα οποία θέλουν ότι είναι σε κίνδυνο μη συμμόρφωση ε, φέτο. Έξι σε σχέση με 8-5 και έξι κράτη-μέλη ε, συνάδουν με το σύμφωνο αυτό σταθερότητα Γερμανία, Γαλλία, ε, Γερμανία, Ολλανδία, Λετωνία και άλλε. Κάποιε θεωρούνται ότι είναι σε γενικέ γραμμέ συνάδουν, η Κύπρος, Μάλτα, Σλοβακία, Εστονία και πέντε άλλα κράτη-μέλη είναι σε κίνδυνο μη συμμόρφωση. Αυστρία, Βέλγιο, Ιταλία, Πορτογαλία και Σλοβενία. Ω εκ τούτου, ζητούμε από όλα τα κράτη-μέλη που είναι σε κίνδυνο μη συμμόρφωση να λάβουν τα απαραίτητα μέτρια στα πλαίσια των εθνικών διαδικασιών, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι ο προπολογισμό του 2018 συνάδει με το EGP και όπω γνωρίζετε αποστήλαμε και μια επιστολή προς τις ε, σχετικές αρχές, ε, προς τον Επιτροπό για να τονίσουμε τη σημασία να ενισχύσουμε τον προϋπολογισμό του 2018 σε ό,τι αφορά τις βασικές διατάξεις τους προκειμένου να μείνει στο επίπεδο διαφορετικών μεταρρυθμίσεων 1,8% για το ΑΕΠ για τις μεταρρυθμίσεις και όπως σας είπαμε Αυτό είναι και μικρότερο ποσοστό από τη δικαιολογή το Μάτρεξ, ο πίνακα. Και τονίσαμε και τη σημασία να συνεχιστούν οι διατροφικέ μεταρρυθμίσει σε ό,τι αφορά τι συντάξει, συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τα. σε ό,τι αφορά και τα κριτήρια χρέωση στην άνοιξη του 2018. Άρα συνολικά διαπιστώνουμε ότι η δημοσιονομική κατάσταση στην Ευρωζώνη σταδιακά βελτιώνεται όλο και πιο λίγες χώρες βρίσκονται σε ε, διαδικασία υπερβολικής ε, χρέωσης, σε κάποιες χώρες είναι σε κίνδυνο ε, μη συμμόρφωσης και σε κάποιες άλλες χώρες διαπιστώνουμε σαφώς μείωση του χρέωση και του ελλείμματος. Και θα δώσω το λόγο λοιπόν στον Πιέρ για να μας εξηγήσει τις αποφάσεις που ελήφθησαν σε ό,τι αφορά το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ευχαριστώ πολύ και το λόγο έχει ο Επιτροπός Μισκοβησή. Ευχαριστώ. Για σε ό,τι αφορά τα οριζόντια ζητήματα που εξετάζουμε σε αυτό το δημοσιονομικό πακέτο, υπάρχει μία διαπίστωση ότι παραμένουν ε, σημαντικέ ε, διαφορέ μεταξύ των μελών. Να ακολουθούμε λοιπόν μια διαφοροποιημένη μελων ακολουθουμε λοιπον μια διαφοροποιημενη προσεγγιση για να υπάρχει ισορροπία μεταξύ ε, τη δημοσιονομική στήριξη και των μέτρων και των προσπαθειών για να διασφαλίσουμε την δημοσιονομική σταθερότητα και βιωσιμότητα. Ε, αρκετή επιτυχία λοιπόν μέχρι τώρα. Θέλουμε να προωθήσουμε μια ευφυή εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητα και Ανάπτυξη. Ε, δηλαδή θέλουμε να τηρήσουμε του κανόνε στο σύνολό του. Και βλέπουμε ότι το μέσο επίπεδο λύματος παραμένει στο 1,1% και 0,9% το 2018. Βλέπουμε ότι κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε το τέλος ε, της ε, διαδικασίας ε, υπερβολικού το 2018. ταυτόχρονα όμως έχουμε και προβληψιμότητα, μάλλον ευελιξία σε, κάποια, σε κάποιες περιπτώσεις, 18% και όχι 19% όπως είπαμε προηγουμένως, γιατί η Ελλάδα παραμένει σε διαφορετική κατηγορία. Η Γερμανία και η Αυστρία έχουν παρουσιάσει δημοσιονομικά προβλέψει ε, σε μια βάση ε, ιδίων πολιτικών και η Ασπανία τελικά υπέβαλε ένα προσχέδιο προπολογισμού με ίδιες πολιτικές ε, εξαιτία μια καθυστέρηση ό,τι αφορά την δημοσιονομική της πολιτική. Όταν θα έχουμε λοιπόν ένα νέο προσχέδιο προπολογισμού. Θα τα επαναξετάσουμε όλα αυτά. Επιστρέφουμε τώρα στην ουσία των γνωμοδοτήσεων. Οι κανόνε ξέρετε ότι ενδιαφέρουν ανάλογα με το κατά πόσο μια χώρα βρίσκεται ε, στο προληπτικό ή διορθωτικό σκέλος ε, του συμφώνου. Αυτοί που έχουν δηλαδή κατά από 3% βρίσκονται στο προληπτικό και έτσι πρέπει να ε, προσαρμόσουν την πορεία τους πρόθεσμα. Πρέπει να διαμορφήσουν λοιπόν ένα περιθώριο ασφαλείας και έτσι να περιορίσουν τους κινδύνους για τα δημόσια οικονομικά και τη βιωσιμότητά τους. Και έτσι πρέπει να τηρείται το κριτήριο του, ε, του χρέους. Οι χώρε τώρα που βρίσκονται στο διορθωτικό σκέλο, πάνω από 3% πρέπει να ε, συμμορφωθούν με τι απαιτήσει του Συμβουλίου και έτσι να μείνουν κάτω από 3%. Καμία χώρα δεν ε, θεωρείται ότι δεν συμμορφούνται ή δεν είναι εντάξει αυτή η κατηγορία της σημαντικής ε, και σοβαρής μη συμμόρφωσης και έτσι δεν έχει ζητήσει και σοβαρή μη αναθεώρηση προσχεδίου προπολογισμού. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι προβληματισμοί σε ορισμένου προπολογισμού. Γι' αυτό έχουμε, και έχουμε ζητήσει επιπλέον στοιχεία από το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Πορτογαλία. Ε, και έχουν ληφθεί όλα αυτά υπόψη και στην ανάλυση μα. Θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η δημοσιονομική προσαρμογή που, ε, ε, που προβλέπεται είναι πέραν των όσων ε, απαιτείται από το Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη. Τώρα να επισέλθω στι λεπτομέρειε, ξεκινώντα από τα 16 κράτη-μέλη στο προληπτικό τμήμα. Έξι χώρε έχουν ε, υποβάλει σχέδιο προπολογισμού που θεωρούμε ότι συμμορφούνται. Ε, πέντε χώρε ε, θεωρούμε ότι κατά σε γενικό βαθμό ε, συμμορφούνται και σε πέντε χώρες ε, υπάρχει κίνδυνος μη συμμόρφωσης με το ε, σύμφωνο για το 2018 σε ό,τι αφορά ιδίω το 0,5% του ΑΕΠ ή 0,25% στα δύο χρόνια. Στο Βέλγιο και την Ιταλία λοιπόν υπάρχει κίνδυνο μη συμμόρφωση σε ό,τι αφορά το κριτήριο τη μειώση του χρέου. Στην περίπτωση τη Ιταλία υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα σχετικά με τι δημοσιονομικέ ε, προβλέψει και τον τελικό προπολογισμό. Έχουμε λοιπόν αποστείλει επιστολή στι Ιταλικές ε, αρχέ για να μα ενημερώσουν για την προθέσει του ό,τι αφορά την επανεξέταση του, της του κριτηρίου της μείωσης του, δανει, του χρέους ε, στην άνοιξη του 2018. Θεωρούμε λοιπόν ότι μια διεθνική προσαρμογή ε, που αποκλίνει από ε, τον μέσο όρο είναι κάτι το αποδεκτό για αυτές τις δύο χώρες. Οι δύο χώρες ε, στην Ευρωζώνη ακόμα υπόκειται στη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος. Για τη Γαλλία λοιπόν θεωρούμε ως σημείο βάσης ότι θα έχουμε κάτω από το 2017. Οπότε εξετάσαμε το σχέδιο του προλογισμού του 2018 ε, υπό το προληπτικό σκέλος. Βάσει τη ανάλυσης με λοιπόν αυτό το προσχέδιο προπολογισμού ε, ενέχει κίνδυνο μη συμμόρφωση με τι απαιτήσει του συμφώνου σε ό,τι αφορά το διασωτικό έλλειμμα. Ε, βλέπουμε ότι υπάρχει εξυγίανση, παρότι θεωρούμε ότι υπάρχει απόκληση σχέση με το 1,1% που είχε προβλέψει η γαλλική κυβέρνηση. Θα περιοριστεί αυτό, αυτό συμβαίνει κάθε χώρο, κάθε χρόνο. Βλέπουμε όμως ότι υπάρχει ακόμα τέτοια απόκληση και μη τήρηση του κριτηρίου της μείωσης του ε, χρέους του 2018 για την Ισπανία. Θεωρείται ότι σφαιρικά συμμορφούνται με τις απαιτήσεις του Συμφώνου του 2018, καθώς οι προβλέψεις του φθινοπόρου του 2017 της Επιτροπής προέβλεπε ε, ονομαστικό έλλειμμα κάτω από το 3% του ΑΕΠ του 2018. Όμως... Ε, ε, έχουμε και αυξήσει ό,τι αφορά τους αριθμούς ε, των μεταναστών και υπάρχουν και δαπάνες ε, για την ασφάλεια, οπότε η Αυστρία έχει ζητήσει επιπλέον ευελιξία του 2017. Συνεχίζεται αυτή η συζήτηση που είναι εξαιρετικά σημαντική για την Ευρωζώνη, παραμένει προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγώ μαζί με τον Βάλτης Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Ξεκινάμε με τις ερωτήσεις. Ο κύριος Χέις για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας καλωσορίζω και τους δύο στη συνεδρία της Επιτροπής ΕΚΟΝ. Έχει υπάρξει αρκετή πρόοδος τα τελευταία χρόνια στον τομέα του χρέους και των ελλημάτων. Κάποιες ερωτήσεις για την Ιρλανδία. Στην Ιρλανδία έχει στη χώρα μου σημειωθεί εξαιρετική πρόοδος τα τελευταία χρόνια μεν, αλλά θα ήθελα να δούμε λίγο το Brexit και πώς ένα σκληρό Brexit μπορεί να επηρεάσει την Ιρλανδική οικονομία. Ε, ξέρω ότι στην πρόταση προϋπαλογισμού που δόθηκε από την Ιρλανδία αναφέρεται στο θέμα αυτό και πώς μπορεί να υπάρξει ένα συμμετρικό σοκ ε, σε σχέση με τις πιθανότητες μείωσης των ρυθμών ανάπτυξης. Ε, τι μορφή μπορεί να έχει ένα τέτοιο ασυμμετρικό σοκ γιατί Νομίζω ότι οι διαπραγματεύσεις μπορεί να μην πάνε καλά, οπότε αυτό το σενάριο δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Τώρα το λεγόμενο output gap στο οποίο αναφέρεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, τετραετής διάρκειας ελέγχου οι οποίες όμως μπορεί να αλλάζουν από τον ένα χρόνο στον άλλο και δεν ξέρω μπορεί να υπάρξει ε, μια αντικειμενική περιγραφή του λεγόμενου output gap ε, και ειδικά για τη δική μου χώρα όπου υπάρχουν πάρα πολλές αλλαγές ε, έχουμε να κάνουμε με μια οικονομία η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλές εξαγωγικές δραστηριότητες όπως επίσης και μια κοινωνία που χαρακτηρίζεται από σοβαρές δημογραφικές αλλαγές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν σε σχέση με τα output gap μπορεί να μας δώσει κάποιες περισσότερες πληροφορίες. Και τώρα για τις αποστολές ελέγχου στο Δουβλίνο. Εμείς φυσικά θέλουμε να βλέπουμε τον κύριο Μοσκόβηση στο Λονδίνο και είναι καλοδεχούμενος. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να τερματίζεται αυτό το πρόγραμμα της εγκύτερης μορφής εποπτείας ε, ιδιαίτερα από του χρόνου όπου θα έχουμε ένα ισορροπημένο προϋπολογισμό οπότε διαρωτώμε αν θα σταματήσουν αυτού του τύπου οι έλεγχοι και μια τελική θα έλεγα παρατήρηση για το επενδυτικό έλλειμμα μήπως μπορούμε να φανταστούμε μεγαλύτερη ευελιξία ε, για τις χώρες που βγαίνουν από πρόγραμμα ε, ποια είναι η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση ε, με τις μεγαλύτερες ευελιξίες στον τομέα των επενδύσεων στις χώρες που λόγω της κρίσης ε, σημείωσαν τρομακτικές μειώσεις στην επενδυτική προσφορά. Ευχαριστώ. Ο κ. Ντομπρόσκης, σας ευχαριστώ για την ερωτήση σας, τις ερωτήσεις σας για την Ιρλανδική οικονομία. Πράγματι η Ιρλανδική οικονομία πηγαίνει πάρα πολύ καλά. 4,8 ρυθμός ανάπτυξης φέτος και αντίστοιχα για του χρόνου. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό το λαμβάνουμε υπόψη μας και σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις με το Brexit παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς τις διαπραγματεύσεις όπως γνωρίζετε δεν έχει υπάρξει αυτή τη στιγμή ένα δεδομένο σενάριο κατάληξης των διαπραγματεύσεων. Πιστεύουμε ότι θα υπάρξει πάντως μια συμφωνία και ένα διατεταγμένο σε εισαγωγικά Brexit. Για το output gap πράγματι έχουμε μια ομάδα εργασίας γύρω από το θέμα αυτό που εξετάζει εξετάζει τους τρόπους τροποποίησης της κοινή μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται στα διάφορα κράτη-μέλη. Απαιτείται η συμφωνία συνεπώς των κρατών μελών για η αδίποτε μορφή αλλαγής. Βλέπουμε ότι κάτι τέτοιο μερικές φορές είναι δύσκολο να γίνει γιατί ορισμένες χώρες αμφισβητούν κάποια τμήματα της μεθοδολογίας, κάποιες άλλες άλλα. Πάντως όταν προσπαθούμε να αξιολογήσουμε το λεγόμενο output gap χρησιμοποιούμε τα μέσα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας για να αξιολογήσουμε ε, τα output gaps των κρατών μελών. Βλέπουμε ότι ε, σε σχέση ε, με τις μεγάλες χώρες οι μικρότερες είναι πολύ πιο πτυτικές σε εισαγωγικά και υπάρχουν μεγαλύτερες διακυμάνσεις στα αποτελέσματα. Και υπάρχει εδώ φυσικά και το θέμα του χρέους το οποίο το παρακολουθούμε από κοντά και στα πλαίσια των προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει το ΔΕΛΤΑ Τώρα για τις ελλείψεις στις επενδύσεις. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε μέσω των ευρωπαϊκών πολιτικών. Αν δείτε την έκθεσή μας για την ετήσια ανάπτυξη, έχουμε συγκεκριμένες ρήτρε για τις επενδύσεις. Το ίδιο ισχύει και με τη ρήτρα στα πλαίσια του Συμφώνου Ανάπτυξης και Σταθερότητας. Και επίσης στα πλαίσια των συστάσεων αναχώρα εξετάζουμε την σύνθεση ε, των τμήματων των προϋπολογισμών των κρατών μελών και σε σχέση με τις επενδύσεις. Υπάρχουν ε, λοιπόν μέσα για την αξιολόγηση ακριβώς ε, των ελλείψεων στον τομέα των επενδύσεων. Θα είμαι σύντομος, ο Βάλντης είπε τα βασικά. Να πω ότι πάντα όταν έρχομαι στην Ιρλανδία είμαι ε, ε, ιδιαίτερα ικανοποιημένος και όταν έρχομαι εκεί τις πιο πολλές φορές συζητώ φορολογικά θέματα παρά τέτοιου θέματα στα οποία εσείς αναφερθήκατε. Και είναι σημαντικός ο ρόλος τον οποίο παίζει η Ιρλανδία σε σχέση με τις αποφάσεις τις οποίες ε, παίρνουμε στον τομέα ας πούμε της ε, μαύρης λίστας των φορολογικών παραδείσων δηλαδή και άλλα θέματα ε, για, την την ενιαία επίσης φορολογική βάση για τις μικρομεσαίες είναι λοιπόν μια καλή ευκαιρία για μένα όταν έρχομαι στο Δοβλίνο και δίνω τις δυνατότητες να σημειώνεται με χαρά ε, τα αρνητικά στοιχεία των πολιτικών προτάσεων τις οποίες κάνουν. Νομίζω ότι ο Βάλτης αναφέρθηκε στους κανόνες οι οποίοι ισχύουν. Αυτή τη στιγμή δεν έχει επιστραφεί το 75% του χρέους. Πρέπει ο κανόνας να γίνεται σεβαστός λοιπόν και εφόσον ο κανόνας ισχύει και μπορεί κανείς να θέσει ερωτήματα σε σχέση αλλά νομίζω ότι οι επιδόσεις σας δεν είναι ε, κακές της χώρας. 5,1 ανάπτυξη το 16 και προβλέπετε 3,9 το 18. Είναι μία από τις ηγέτιδες χώρες σε επίπεδο ρυθμών ανάπτυξης και αυτό το σημειώνουμε με πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα ήθελα να πω ότι κάναμε και μια αποστολή επιτυχέστατη πρόσφατα στην Ιρλανδία και είδαμε τα πράγματα και δεν έχουμε νομίζω κάτι να φοβηθούμε και όταν τα πράγματα επιταχυνθούν ακόμα περισσότερο το πρόγραμμα αυτό ε, ελέγχου αν θέλετε σε επίπεδο εγκύτερο θα διακοπεί. Τώρα για το Brexit. Ε, προς το παρόν ε, οι αρνητικές επιπτώσεις ε, περιορίζονται στις συνέπειες της μείωσης της ισχύω της στερλίνας και κάποιες αυξήσεις τιμών για τους Ιρλανδούς καταναλωτές. Οι προβλέψεις μας για το 18 βασίζονται σε εντελώς τεχνικές αν θέλετε διαπιστώσεις ε, ε, διατήρησης του status quo ε, ανάμεσα στις 27 χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο. Και αυτό δεν έχει κάποια σχέση με το άρθρο 15 της συνθήκης. Αυτό το κάνουμε λαμβάνοντας μέτρα τα οποία δεν συνιστούν μια πολιτική θέση. Είναι μια, μια ανοιχτή χώρα η Ιρλανδία με πάρα πολλές ε, ε, μεγάλες επιχειρήσεις, πολυεθνικές επιχειρήσεις και με πολύ στενές σχέσεις και με άλλες χώρες όπως οι Ενωμένε Πολιτείες. Τώρα για την ενιοποιημένη φορολογική βάση νομίζω ότι το CCCTB θα το υιοθετήσουμε πάρα πολύ σύντομα από κοινού όλοι. Θα ομιλήσω την Πορτιγαλική λέει ο κύριος Περέιρα. Δύο ερωτήσεις να σας κάνω. Η πρώτη. Μία πιο γενική. Αξιολογώντας τα προσχέδια προϋπολογισμού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει σε συζητήσει με τα κράτη-μέλη όχι μόνο σε ό,τι αφορά τη συμμορφωσή του με του κανόνε, αλλά και για την ερμηνεία των κανόνων. Σε κάποιε περιπτώσει υπάρχουν σημαντικέ αποκλήσει, σημαντικέ αποκλήσει σε ό,τι αφορά την ερμηνεία, σε ό,τι αφορά το δυναμικό κινδύνου, το δυναμικό ανάπτυξη για το διορθωτικό έλλειμμα και το ίδιο διαπιστώνουμε και με όρους όπως η κατατάξη των έκτακτων μέτρων, οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες, η Eurostat. Σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζονται μήνες ολόκληρους για το πώς θα κατατάξουν το εκάστοτε μέτρο. οι κανόνες για τον προϋπολογισμό. Φαίνεται ότι έχει καταστεί πολύ σκοτεινή υπόθεση και κανείς δεν φαίνεται να τον λαμβάνεται αυτό πλήρω. Πώς μπορείτε λοιπόν να ανταποκριθείτε, ρωτώ αγαπητή Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις εκκλήσεις των κρατών μελών να διευκρινιστούν σε κάποιες περιπτώσεις ε, οι κανόνες. Δεύτερη ερώτηση σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα την Πορτογαλία. Παρά τους κινδύνους τους οποίους έχει εντοπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όλοι να γνωρίζουν, όλοι συμπεριλαμβανομένοι και της Επιτροπής, ότι η δημοσιονομική κατάσταση στην Πορτογαλία βελτιώνεται. Βελτιώθηκε μάλιστα σημαντικά το φετινό έτος. Η χώρα αναμένεται ότι θα αυξηθεί φέτος με πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από το ευρωπαϊκό μεσόωρο. Πάνω από το ευρωπαϊκό λοιπόν μεσόρο και μειώνεται και τις προβλέψεις σας για τη χρέωση και το δημόσιο έλλειμμα. Το 2015 μιλούσαμε για επιδείνωση του δημοσίου ελλείμματος, για κυρώσεις ενδεχομένω. Σήμερα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί ότι υπάρχει μείωση του ελλείμματος το 2016 και το 2017 και το 2018 κατά πάσα πιθανότητα. Το θέμα είναι η κλίμακα μείωσης του δημοσίου ελλείμματος, κατά είναι επαρκή. Και ρωτώ λοιπόν, τα προηγούμενα αποτελέσματα έχουν οδηγήσει σε κάποια θετική επανεκτίμηση των προβλέψεων από το διάλογο με τις πορτογαλικές αρχές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σχηματίσει μια εντύπωση εμπιστοσύνη προς τις πορτογαλικές αρχές και προς την πορτογαλική οικονομία για την δυνατότητα της να συνεχίσει να μας εκπλήσει με τα θετικά αποτελέσματα αυτά. Ευχαριστώ απάντηση. Κοιτάξτε, για τα δύο αυτά σημεία, καταρχά, σε ό,τι αφορά τον διάλογο, υπάρχει τριφωτικό ε, διάλογο και υπάρχουν κοινοί κανόνε και κώδικε και στατιστική κατάταξη για όλα τα θέματα αυτά, σε ό,τι αφορά και την προβλεψιμότητα. Είναι λοιπόν μια εργασία ανεξελίξη σε ό,τι αφορά την πορτογαλική οικονομία τώρα. Θα θυμάστε Υπάρχει εκτίμηση, υπάρχει κρίση ότι είναι η οικονομική της στην Πορτογαλία αρκετά στεναρή. Ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα σαφώς είναι σε μείωση, σε σημαντική μείωση, μειώνοντα σημαντικά. Και κατά τρίτον, ότι γίνονται διαφορετικές προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Όπως όμως αναφέρατε, αυτές οι διαφορετικές προσπάθειες δεν επαρκούν δεν τα δεδομένων των κριτηρίων που ισχύουν. Έπρεπε λοιπόν να το αναφέρουμε αυτό και να ζητήσουμε περαιτέρω προσπάθειες. Αληθεύει επίσης ότι στο παρελθόν έχουμε παρατηρήσει ότι τα αποτελέσματα στην Πορτογαλία ήταν καλύτερα από τι προβλέψεις μας. Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη γιατί προφανώς εμείς πρέπει να κάνουμε μετριοπαθείς προβλέψεις. Πρέπει να δείξουμε ήπια και μετριοπαθή στάση στις προβλέψεις μας. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, προφανώς, προσαρμοζόμαστε. Υπάρχει λοιπόν εμπιστοσύνη προς την πορτογαλική οικονομία. Η απάντησή μου θα ήταν ναι. Η εμπιστοσύνη αυτή δεν ε, διακυβεύει ωστόσο την ανάγκη διαρθωτικών ε, προσαρμογών. Και εκεί προφανώς ε, συνοψίζεται η στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ένα σημείο προσοχής για το μέλλον, γιατί η Πορτογαλία προφανώς είναι σε υψηλή φάση του κύκλου και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να συνεχιστούν οι διορτικές μεταρρυθμίσεις απαρεγκλήτως. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Από την άλλη τώρα, η κυρία Πίκνικ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητέ κυρία Μεντομπρόφη και κύριε Μοσκοβισή, Κατάρχά χαίρομαι με την ελαφριά βελτίωση σε ό,τι αφορά τα σχέδια, τα προσχέδια προπολογισμού. Ένα κράτο λιγότερο κίνδυνο μη συμμόρφωση. Σήμερα θα ήθελα να μιλήσω σε ό,τι αφορά την περιπλοκότητα των τρέχοντων κανόνων. όπω είπε πρώτα του Eurogroup πρόσφατα, σε ό,τι αφορά τους κανόνες του, του ε, Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, οι κανόνες είναι πάρα πολύ εμ, περίπλοκοι. Και προτάθηκε το 2016 απλοποίηση για να, να βασιζόμαστε σε ένα ε, στοιχείο, είτε στο έλλειμμα είτε στο χρέος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει μια τέτοια προσέγγιση για να γίνει επιλογή δηλαδή ε, μεταξύ ενός των δύο αυτών παραγόντων και αν ναι, ποιον θα διάλεγε. Επίσης αναφέρθηκε ότι οι κανόνες είναι περίπλοκοι και θα πρέπει σε κάποια περίπτωση να υπάρχει και ένα ποσοστό ευελιξίας. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό η έκθεση EFB αναφέρει ότι η περιπλοκότητα αυτή θα μπορούσε να μειωθεί με κάποιες ρήτρες διαφυγής. Και έτσι ορίζονται τέσσερις όροι για την κινητοποίηση μια ρήτρα, ε, μάλλον για να μπορεί να υπάρχει αυτή η ρήτρα διαφυγή. Η τρίτη και η τέταρτη θα πρέπει να περιλαμβάνουν ανεξάρτητες αξιολογήσει και συστάσει από ανεξάρτητο σώμα προκειμένου να αποφευθεί η ευκαιριακή και οπορτουνιστική χρήση. Συμφωνείτε με την έκθεση EFB και ποιο πιστεύετε ότι θα πρέπει να διαδραματίσει το ρόλο ανεξάρτητου τέτοιου σώματο. Για παράδειγμα αυτή η ευθύνη θα μπορούσε να είναι της EFB, μιας Γενικής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή ενδεχομένως μιας νέας υπηρεσίας. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Of course we Σας ευχαριστώ και προφανώς εδώ οι συνθήκες ορίζουν τα πράγματα με σαφήνεια. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση αυτή και όντως σε ό,τι αφορά την περιπλοκότητα των κανόνων Αυτό θα πρέπει να το αξιολογήσουμε στην τρέχουσα φάση. Δεν είναι 100% ξεκάθαρα τα πράγματα σε ό,τι αφορά τις συζητήσεις μας. Γιατί αν απλοποιήσουμε υπερβολικά τους ε, κανόνες, ε, συχνά αντιμετωπίζουμε ε, ενστάσεις από τα κράτη-μέλη του. δεν έχει ληφθεί υπόψη το χύψη στοιχείο και δεν αποτυπώνεται η πραγματική κατάσταση. Φυσικά όταν αρχίζει κανείς να λαμβάνει υπόψη πιο πολλού παράγοντες, οι κανόνε καταλήγουν να είναι πάρα πολύ περιπλοκοί. Άρα υπάρχει, ξέρετε, μια χρυσή τομή η οποία θα πρέπει να βρεθεί μεταξύ της περιπλοκότητας και των τρέχουσων τάσεων. Τα μη παρατηρούμενα κριτήρια επίσης, ε, output gap και σε ό,τι αφορά το ισοζύγιο των διαφορετικών αυτών στοιχείων. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να προποιήσουμε τους κανόνες, πώς μπορούμε να τους τα καταστήσουμε πιο προβλέψιμους. Αυτή η δουλειά γίνεται και στο ΕΚΟΦΗΝ άλλωστε. Έγινε το ΕΚΟΦΗΝ υπό Ολλανδική Προεδρία στο Άμστερνταμ και φαίνεται ότι υπάρχει μια κάποια σύγκληση για να, να υπάρχουν πιο πολλά ορόσημα δαπανών, benchmarks δαπανών. Έχουμε λοιπόν ελέγχο των δαπανών καταρχάς και ε, σε ό,τι αφορά τη μεγαλύτερη περίοδο ομαδοποίησης για να μειωθεί η διακύμανση. Αυτό πλέον χρησιμοποιείται στο, στις Σε ό,τι αφορά το έλλειμμα και το χρέος, θα έλεγα ότι και τα δύο κριτήρια πρέπει να ακολουθούνται γιατί σε μακροπρόθεσμα μεγαλύτερη χρονική περίοδο μπορούσε, θα προτιμούσε κανείς να προτιμήσει το κριτήριο της χρέωσης γιατί αυτό προφανώς έχει μεγαλύτερη επιρροή στη βιωσιμότητα των δημοσιονομικών αλλά αυτό που είναι πιο εύκαιρο για τους πολιτικούς ανά πάσα στιγμή είναι το έλλειμμα και όχι το χρέος. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να λεφθεί υπόψη. Σε ό,τι αφορά την ευελιξία τώρα, Υπάρχει μια κάποια ευελιξία στο Σύμφωνο Θεραπευτές και Ανάπτυξης. Αυτή η ευελιξία λοιπόν ήδη αποτυπώθηκε σε ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βέλτιστη χρήση της ευελιξίας σε ό,τι αφορά τους κανόνες του Συμφώνου Θεραπευτές και Ανάπτυξης, το πώς ε, χρησιμοποιούνται οι ρήτρες ε, ε, και τη μεταρρύθμιση κτλ. και πώς όλα αυτά εντάσσονται στον οικονομικό κύκλο. Και στο σημείο λοιπόν αυτό γίνεται κάποια αξιολόγηση και εκτίμηση. Δεν εφαρμόζονται όλα με αυστηρούς μαθηματικούς ε, τρόπους. Επίσης, λαμβάνεται υπόψη το σκέλος της επιτήρησης της οικονομικής απόδοσης των κρατών μελών από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πιστεύουμε ότι αυτό θα πρέπει να παραμείνει έτσι. Και προσφάτως είπαμε ότι το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό, η Ευρωπαϊκή Δημοσιονομική Επιτροπή δίνει ανεξάρτητες συστάσεις και εξπόστ την εφαρμογή των κανόνων και συστάσεις εξάντεκ προτέρων για την σωστή δημοσιονομική στάση και η σύσταση του τελευταίας ε, έκτασης της Επιτροπής αυτής ήταν ότι συνολικά ήταν ικανοποιητική η εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Δεν ε, ήταν αυστηρή αυστηρότατη, αλλά υπήρξε μια εξισορρόπηση μεταξύ δημοσιονομικής βιζιτιμότητας και οικονομικής ανάπτυξης και των αντίστοιχων αναγκών που επικρατούν σε κάθε οικονομία. Ευχαριστώ. από την παρακαλώ. Θα μιλήσω πρωτογαλλικά. Δύο ερωτήματα. Πρώτον, για τη μεθοδολογία και ένα δεύτερο πιο γενικό ερώτημα. Στην εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το προσχέδιο προπολογισμού της Πορτογαλίας γίνεται λόγος για δεκα... διψήφια ποσοστά. Αν υπολογίσετε το πιθανό ΑΕΠ, το οποίο βέβαια αντανακλά και τις ε, διαθετικές ισορροπίες και τις ε, δαπάνες, νομίζω ότι η στόχη είναι πολύ κοντά. Και πρόκειται για ιδιαίτερα μετάβλητα μέτρα. Οπότε, γιατί θεωρείτε ότι η Πορτογαλία βρίσκεται σε κίνδυνο μη συμμόρφωση για τον πληθυσμό, για, για τους Πορτογάλους πολίτες. Είναι δύσκολο να κατανοήσουν, γιατί όταν έχουν ένα ονομαστικό έλλειμμα 1,4% ε, θεωρείται ότι διατρέχουν κίνδυνο μη συμμόρφωση. Και μάλιστα σε μια χρονική στιγμή που οι Πορτογάλοι έχουν κουραστεί από αυτή την αίσθηση της καταδίωξης και της, ε, και της εκβιαστικής προσέγγισης από πλευράς Κομισιόν εδώ και πολλά χρόνια. Ένα δεύτερο πιο γενικό ερώτημα. Η Πορτογαλία από το 2015 ακολουθεί μια νέα τροχιά αποκατάστασης ε, των, ε, των απολαβών εργαζομένων και στεξιούχων. Όμως στην Πορτογαλία έχουμε ακόμα εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους με μισθούς και συντάξεις 200-300 ευρώ το μήνα. Απαιτείται λοιπόν ε, διεύρυνση των δαπανών, αλλά αυτό βέβαια έχει να κάνει μετά και με το ισοζύγιο. Το 0,25% ε, πλεόνασμα είναι ο ενδιάμεσος στόχος, δεν είναι υπερβολικός για μια διαθετική τέτοια ισορροπία, για μια χώρα όπως η Πορτογαλία, που ακόμα έχει να κάνει με πολλές ε, ανεπάρκειες, δυσλειτουργίες, ελλείψεις δημοσίων ταπανών. Ο μεσοπρόθεσμος στόχος να θεωρείται λίγο υπερβολικός. Ε, δεν θα αναθεωρήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτόν τον στόχο. για να φύγουμε από τον δρόμο της λιτότητας. Ε, Κύριε Βιέγκας, αρχικά θα ήθελα να υπενθυμίσω τους κανόνες μας. Γιατί εμείς ε, τους κανόνες ακολουθούμε. Δεν τους επινοούμε, απλώς τους εφαρμόζουμε. Εάν εξετάσουμε λοιπόν και τους ε, κανόνες ε, δαπανών ε, και τα ελλείμματα, πράγματι προβλέπεται σημαντικό, κίνδυνο σημαντικής απόκλησης σε σχέση με τα απαιτούμενα επίπεδα που είναι το 0,6% και το 17% και το 18%. Το ανέφερε και στον κύριο Περέιρα ότι αυτό βέβαια δεν μας εμποδίζει να θεωρούμε ότι οι προσπάθειες που έχουν καταβληθεί δεν είναι αμελητές, το κάθε άλλο και ε, κάποιες φορές αυτές ε, οι αποκλήσεις διορθώνονται ε, μέσα στη χρονιά, αυτό το έχουμε δει στο παρελθόν, οπότε έχουμε εμπιστοσύνη στην πορτογαλική οικονομία, είναι και μια χώρα που ξέρω καλά. Μια άλλη μάλλον χώρα που γνωρίζω καλά και επίσης αυτή αντιμετώπιζε τα ίδια ζητήματα είναι η Γαλλία, αλλά βλέπουμε ότι, με μεγάλη χαρά, ότι αυτή η χώρα μπορεί να φύγει από την διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος. Οπότε και οι λέξεις έχουν το νόημά τους, αλλά είναι μια διαδικασία που δεν έχει άμεση επιπτώσει. Απλώ ε, ξεκινάει ένα επικοδηματικό διάλογο που κάνουμε τώρα αυτή τη στιγμή με την πορτογαλική κυβέρνηση. Ε, δεν χρειάζεται λοιπόν ε, να το περιβάλλουμε όλο αυτό με συναισθηματισμούς που αυτή τη στιγμή δεν χρειάζονται. Εμείς πράγμα μαζί. Τώρα, σε ό,τι αφορά γενικά την πορτογαλική οικονομία, Βεβαίω δεν μπορούμε να παρέμβουμε στα εσωτερικά της Πορτογαλίας. Μια χώρα ε, με ιδιαιτερότητες και πλούσιο και ζωντανό πολιτικό διάλογο. Μου φαίνεται ότι αυτά που είπατε εσείς για μια νεοφιλελεύθερη πολιτική που θέλει να επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, νομίζω ότι δεν ισχύουν για αυτή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνήθηκε όταν η Πορτογαλία είχε κάνει τις ε, προσπάθειες για να φύγει από το πρόγραμμά της, αρνήθηκε λοιπόν να επιβάλλει πολιτική λιτότητα στην Πορτογαλία. Εμείς ε, δεν επιβάλλουμε τίποτα ε, στις Επιμέρου κυβερνήσει και στην τωρινή και στην προηγούμενη να ακολουθήσει ε, δημοσιονομικέ πολιτικές. Εγώ χαίρομαι μάλιστα που αυτή η πολιτική που ακολουθείται δεν είναι νεοφιλελεύθερη. Οπότε δεν θέλουμε να επιβάλλουμε τίποτα στην Πορτογαλία. Και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κατάλοιπα της κρίσης, υπάρχουν ανισότητες και δυσκολίες που τις ε, βιώνουν πολλοί συμπολίτε σας. Εμείς πάντα θέλουμε να εφαρμόσουμε τους κανόνες, πάντα όμως έχοντας υπόψη και την κατάσταση και ξέρουμε ότι δεν ακολουθούμε τυφλά τους κανόνες. Πράγματι υπήρχε και μια τέτοια συζήτηση το καλοκαίρι του 2016, όπου σκεφτόμασταν αν θα επιβάλλουμε ε, πρόστιμα στην ε, Πορτογαλία αλλά νομίζω ότι πολύ σωστά θεωρήσαμε ότι δεν ε, ε, χρειαζόταν εκείνη τη στιγμή και ότι έπρεπε να περιμένουμε και όντω καλά κάναμε γιατί ένα εξάμεινο αργότερα βγήκε από την όλη διαδικασία Πορτογαλία. Οπότε δεν πρέπει να αμφιβάλλετε για τι καλέ προθέσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και για τους μεσοπρόθεσμους ε, στόχους που ανέφερα, νομίζω ότι σας απάντησα, λέει ο Επίτροπος αδιαπραγμάτευτη. Οι κανόνες ε, βλέπετε λοιπόν ένα έλλειμμα 0,5%. Θα μπορούσε να τροποποιηθεί αν υπήρχε κυκλικά μια αρνητική ε, επίδοση, το οποίο ευτυχώς δεν ισχύει. Νομίζω ότι τα πηγαίνετε πολύ καλά, οπότε δεν χρειάζεται παραπάνω. Ευχαριστούμε. Για τα εγγραφικά ταμεία το Κοινοβούλιο συνσέφερε σε αυτή την ε, σοφή απόφαση. Είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση πράγματα γιατί ε, πράγματι ο στόχος είναι 0,1% μέχρι 0,1%. δεν είναι ρόλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θέσει το NPO. Ε, τα κράτη-μέλη το αναλαμβάνουν αυτό. Βέβαια και η Επιτροπή έχει ε, την δική της εκτίμηση για την ε, διαδικασία. Μάρκο Βάλλη, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις η πρώτη ίσως να αναφέρεται περισσότερο στο προηγούμενο πάνελ, αλλά δεν είχα το λόγο. Θα ήθελα να μου πούνε οι δύο επίτροποι για τα θέματα των ελλημάτων, αλλά κυρίως για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες και για χώρες όπως η Ολλανδία και η Γερμανία. Πότε θα προσπαθήσετε να αναζητήσετε λύσεις των προβλημάτων στον χώρο αυτό. ιδιαίτερα στα πλαίσια της αναθεώρησης του ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου για τις πιθανές χρήσεις των πλεονασμάτων των χωρών αυτών. Και τι θα γίνει με τα χρέη χωρών όπως η δική μου σε πολύ υψηλό επίπεδο μια μικρή μείωση, διορθωτική θα έλεγα, όπως ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε ποιο βαθμό μπορεί να βοηθήσει τα πράγματα. Μήπως θα πρέπει να προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα που έχουμε με καλύτερο τρόπο και μήπως θα πρέπει να δαπανίσουμε σήμερα ε, για να μειώσουμε επί της ουσίας το χρέος και όχι να προσπαθούμε μόνο με φορολογικές παρεμβάσεις ε, να μειώνουμε το κόστος τους. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας, για τις μακροοικονομικές ανισότητες, τις διαδικασίες αυτές. Πράγματι το συζητήσαμε το θέμα αυτό στην προηγούμενο γύρο των συζητήσεων και αυτό το οποίο βλέπουμε είναι κάποιες μακροοικονομικές ανισότητες όχι μόνο στα πλαίσια των ελλημάτων αλλά και των μεγάλων πλεονασμάτων. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο η Ολλανδία και η Γερμανία έχουν μπει στη διαδικασία ακριβώς μακροοικονομικών ανισορροπιών. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εξετάζεται από πλευράς του μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό στην επόμενη έκθεσή μας και στα πλαίσια επίσης και των ειδικών αναχώρα εκθέσεων σχετικά με τις χώρες αυτές. Ε, τώρα, για την ε, δημοσιονομική αν θέλετε πορεία και για χώρες όπως ε, η Ιταλία ε, η αξιολόγηση την οποία κάνουμε είναι ότι θα πρέπει να εξισορροπηθεί η ανάγκη για την οικονομική ανάπτυξη από τη μία με την δημοσιονομική βιωσιμότητα από την άλλη. Και στα πλαίσια αυτά οι χώρες οι οποίες έχουν υψηλά επίπεδα χρέους και υψηλές ανησυχίες κατά συνέπειας για τη βιωσιμότητα των δημοσιονομικών τους θα πρέπει να συνεχίσουν τις διαδικασίες ε, μεταρρυθμίσεων έτσι ώστε να βελτιώσουν ε, την κατάσταση. Έχετε υψηλότατα επίπεδα χρέους ε, μετά την Ελλάδα το υψηλότερο σχεδόν και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξουν ρυθμίσεις έτσι ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση και να είμαστε σε θέση να αποφύγουμε και να αντιμετωπίσουμε μάλλον καλύτερα κάποια μελλοντικά αρνητικά συμβάντα. Άνεμαντς. Ευχαριστώ πρόεδρε και θα μιλήσω Ολλανδικά. Θα ήθελα να συζητήσω με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το σχέδιο προπολογισμού του Βελγίου. ο Γιώργο Παπαδόπουλο, Υπουργός Οικονομικών, αναφέρεται στην ε, δύναμη της αλλαγής για τη μείωση του χρέους, για την εξασφάλιση των μελλοντικών γενναιών. Παρά τις ε, μεγάλες προλογικές ε, προσπάθειες των τελευταίων χρόνων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώνει ότι αυξάνεται η χρέωση του Βελγίου και ότι το, μάλλον ότι το έλλειμμα συνεχίζει να αυξάνεται και ότι η χρέωση σημειώνεται πολύ ε, λιγότερα από ό,τι θα έπρεπε. Μπορείτε να κάνετε μια πιο εντελεχή ανάλυση σε ό,τι αφορά την χρέωση του Βελγίου και τους κινδύνους με προθεσμό επίπεδο θα μπορούσατε να τις περιγράψετε σε ό,τι αφορά το risk, το κίνδυνο σημαντική απόκληση από, το, από την οδό των μεταρρυθμίσεων για τη μείωση του ελλείμματος. Μου φαίνεται πάρα πολύ σοβαρό αυτό ως φαινόμενο και θα ήθελα να καταλάβω αν είναι όντως τόσο σοβαρό όσο ακούγεται. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά το Βέλγιο, η κατάσταση σαφώς βελτιώνεται σύμφωνα και με τις προβλέψεις μας Πιστεύουμε ότι από 2,5% το έλλειμμα θα πάει στο 1,5% το 2017 και σε διαφορετικού όρους περιμένουμε από βελτίωση 0,7% σε σχέση με το ΑΕΠ Είναι λοιπόν πολύ σαφής και θετική τάση. Έχουμε και διάλογο με την κυβέρνηση και τώρα πραγματικά πετυχαίνουμε αποτελέσματα. Και του τουλεχθέντους έχουμε δύο ανησυχίες σε ό,τι αφορά την πρόοδο που έγινε το 16 17 από κοινού δεδομένης της σημαντικής απόκληση από το, το δημοσιονομική του ε, κανόνα του 2017 αναμένουμε ότι από κοινού θα ξεπεραστούν τα περιθώρια και η απόκληση του Βελγίου είναι οριακή σε ό,τι αφορά το 2018 και το 2016-2017 ήταν υπερβολική. Επιβεβαιώνεται λοιπόν αυτό ο κίνδυνο και γι' αυτό καλούμε τι άρχε να καταβάλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου στον προπολογισμό του 2018 να υπάρχει συμμόρφωση με του κανόνε και έχουμε την, την εντύπωση ότι η διαβούλευση, μάλλον η ανάπτυξη στο Βέλγιο έχει να κάνει με τι δαπάνε. Αυτέ είναι προβλέψει για τη βελτίωση τη κατάσταση, αλλά ακόμα θα πρέπει να πετύχουμε και περαιτέρω πρόοδο. Από ό,τι καταλαβαίνω, πρόεδρε, για να ευκρινίσω. Τρία λεπτά, τρία λεπτά μήχα Εξίσου καταλαβαίνω ότι καλά πάνε τα πράγματα. Δεν είσαστε και σε κατάσταση πανικού. Και το 105% του ΑΕΠ θεωρείται θα το πετύχουμε σύμφωνα με τις ε, προβλέψεις σας σε ό,τι αφορά και την έκθεση που έχουμε μπροστά μας. Ναι, νομίζω ότι είχα απαντήσει στην ερώτηση αυτή, όντω. Thank you, Tom Van Ο κύριος Βαντεκάνελάρα, ευχαριστώ πρόεδρε. Ένα ερώτημα λοιπόν για τον Αντιπρόεδρο των Πρόσκης. Βάσει των ε, παραδειγμάτων της Ιταλίας και του Βελγίου, Έχουμε λοιπόν δει ότι δεν πληρούν το κριτήριο του, το benchmark δηλαδή για την μείωση του χρέους και αυτό είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί και για το Βέλγιο γιατί έχει το τρίτο μεγαλύτερο ε, χρέος μετά την ε, Ελλάδα, την Ιταλία και την Πορτογαλία αλλά μετά έχουμε να κάνουμε και με το δεύτερο μεγαλύτερο κόστος γύρανση του πληθυσμού στην Ευρώπη. Μόνο η Σλοβενία ε, έχει χειρότερα στοιχεία. Μέχρι το 2040, όταν θα φτάσει δηλαδή στο απόγειό της γύρανση, ε, τα το κόστος αυτό θα είναι 13 δις παραπάνω σχέση με σήμερα. Οπότε και για το Βέλγιο αλλά και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες η γύρανση ε, είναι το μεγάλο πρόβλημα το οποίο δεν συζητάει κανείς. Όμως εδώ στο, ε, στη δέσμη για το φθινόπωρο, το Atom Package είναι κάτι το οποίο αναφέρεται συγκεκριμένα και είναι πολύ δύσκολο να εξετάσουμε ένα θέμα σαν την γύρανση του πληθυσμού για να το περιγράψουμε με κάθε σαφήνεια και να βρούμε εναλλακτικέ λύσει βράχη και μεσοπρόθεσμα. Δεν ξέρω κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να διδραματίσει χρήσιμο ρόλο εδώ στι συστάσει ό,τι αφορά την γύρανση και τι προβλέψει για τη γύρανση. Με ποιον τρόπο λοιπόν μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, αναλάβει μεγαλύτερο τμήμα αυτής της ευθύνης ε, για να, ε, κάπως, να μετριάσουμε τον αντίκτυπο της γύρανσης του πληθυσμού στην Ευρώπη. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, σε ό,τι αφορά τις δημοσιονομικές επιδόσεις, εμείς ε, ε, παρακολουθούμε τα όσα συμβαίνουν βραχυπρόθεσμα, ε, στις επιδόσεις δηλαδή για το χρέος και τα ελλείμματα. Και κατά μέσο όρο βλέπουμε ότι το έλλειμμα μειώνεται στο Βέλγιο, 2,5% και προβλέπεται 1,5% για φέτος 1,4 του χρόνου. Θεωρούμε λοιπόν ότι η διαφορετική ε, ισορροπία διατηρείται και φέτος και για του χρόνου, όμως η συνολική μας εκτίμηση είναι ότι το Βέλγιο διατρέχει κίνδυνο μη συμμόρφωσης, γιατί βέβαια είναι τέτοια τα επίπεδα δημόσιου χρέους που πρέπει να εξετάσουμε πρέπει να, να δούμε σημαντική μείωση και στο ε, έλλειμμα και ε, στο χρέος. Ωστόσο βλέπουμε ότι ακολουθείται πτωτική τάση και στο χρέος και στο έλλειμμα. ...103,5 φέτος, 102,5 του χρόνου. Ε, επίσης, ε, εκτιμούμε την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών και η γύρανση του πληθυσμού αλλά και οι προεκτάσεις ε, στον ασφαλιστικό κλάδο και ε, στην υγειονομική περίθαλψη είναι κάτι το οποίο εξετάζουμε. Γι' αυτό και συστήνουμε την υιοθέτηση μέτρων σε ό,τι αφορά τι ε, μεταρρυθμίσεις του συνταξιοδοτικού, μεταρρυθμίσεις, μάλλον συντάξεις δεύτερου πυλώνα, για σύνδεση μεταξύ της ηλικίας συνταξιοδότησης και ε, του προσδόκιμου ζωής. Μία σειρά λοιπόν μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι και στην περίπτωση της γύρανσης του πληθυσμού, του πληθυσμού θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την ε, βιωσιμότητα των δημοσίων και αυτό φαίνεται και από την δημοσιονομική ε, μας εξέταση και ανάλυση, αλλά και στις ε, ειδικέ αναχώρες ε, συστάσεις, όπου έχουμε προτάσεις και για την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα. Ευχαριστώ. Okay, so... Καλώς. Σας ευχαριστώ όλους. θα ήθελα να κάνω ένα μικρό σχόλιο. Προσωπικά έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν ειδικέ καταστάσεις σε ορισμένες χώρες, αλλά συνολικά αναγνωρίζουμε την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μπορέσει να εφαρμόσει το σύστημα των κανόνων τα οποία έχουμε με έξυπνο τρόπο, με ευφυή τρόπο στα πλαίσια του οικονομικού κύκλου και σε μια εποχή ανάκαμψης μεν οικονομικής αλλά με χαμηλά επίπεδα αμοιβών και με ελλείψεις στον τομέα των επενδύσεων. Ταυτόχρονα είναι αληθές ότι οι διαδικασίες που θα επιτρέπουν να βελτιωθεί η κατάσταση είναι περίπλοκες και αποδεικνύεται να υπάρχει, ότι υπάρχει και μία κάποια κόποση για την εφαρμογή των ευέλικτων αλλά και πολύ περίπλοκων κανόνων που πρέπει να εφαρμοστούν και όπου έχουμε εφαρμόσει μέχρι τώρα. Απαιτείται μια ολόκληρη σειρά τεκμηρίωσης και συνειδητοποιώ ότι είναι δύσκολο να αλλάξει η κατάσταση αυτή γιατί υπάρχουν ξεκάθαροι κανόνες στη συνθήκη, υπάρχουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις και απαιτείται νέα νομοθετική ε, παρέμβαση για να υπάρξουν αλλαγές αλλά με ενδιαφέρει λίγο να δούμε το πώς μπορείτε να συνδυάσετε τις διαπιστώσεις τις οποίες κάνατε με τα επόμενα βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Πρώτα η διαδικασία συζήτησης για την απλοποίηση και δεύτερον για το τι αναμένετε ότι θα συμβεί ε, με το Fiscal Compact το οποίο από τη μία εάν δεν αναφέρεται στα θέματα της νομοθεσίας αυτό περιορίζεται. Από την άλλη υπάρχουν ορισμένες συνιστώσεις του Fiscal Compact που επηρεάζονται από την συγκυρία. Φυσικά το Κοινοβούλιο θα ήθελε σε αδίποτε νομοθεσία νομοθετική να συμμετέχει πλήρως. αλλά πέραν τούτου αυτό το οποίο με ενδιαφέρει είναι ο τρόπος με τον οποίο εσείς βλέπετε να εξελίσσεται η κατάσταση, η πορεία την οποία ακολουθούμε με βάση τους ισχύοντες κανόνες οι οποίοι όμως ε, δημιουργούν ένα μηχανισμό περίπλοκο που θα πρέπει φυσικά να γίνεται ε, σεβαστός. Άλλωστε εδώ θα ήμασταν πάρα πολύ επιφυλακτικοί εάν ε, υπάρξει ένα συμβούλιο δημοσιονομικό το οποίο δεν καλύπτεται από τους κανόνες και τις προβλέψεις που έχουμε σήμερα. Πάντως θα ήθελα να μάθω με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να έχουμε μέσα και εργαλεία έτσι ώστε να συνδυάσουμε καλύτερα τις εθνικές δημοσιονομικές πολιτικές με τους κοινούς κανόνες και με την οικονομική πραγματικότητα με ισότιμο και αποτελεσματικό τρόπο. Ο κ. Ντομπρόφσκης, σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας Πράγματι και αυτό είναι κάτι το οποίο στην παρούσα φάση συζητάμε. Προσπαθούμε να ισορροπήσουμε ανάμεσα στην απλοποίηση των κανόνων και στην λύπηση υπόψη όλων των παραγόντων που παίζουν ρόλο. Δεν προωθούμε λύσεις υπεραπλούστευσης, γιατί αυτό μπορεί να είναι ελκυστικό σε ένα επίπεδο, από την άλλη όμως όταν εφαρμοστούν σε μια κατάσταση δεν αναγνωρίζουν τις ισχύες της πραγματικότητες. Πρέπει λοιπόν να αποκαταστήσουμε μια κάποια ισορροπία σωστής εφαρμογής των κανόνων από τη μία σωστής προβλεψιμότητας των εξελίξεων από την άλλη. Και όταν μιλάμε για το output gap, έρχομαι σε αυτά τα οποία συζητήθηκαν στο Άμστερνταμ, ε, στο Εκοφίν, σχετικά με τα επίπεδα τα οποία θα πρέπει να ε, πετύχουν τα διάφορα κράτη-μέλη, σχετικά με τα benchmarks τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και ανάλογα και με την περίοδο η οποία κάθε φορά λαμβάνεται υπόψη. Εμείς λοιπόν ε, εργαζόμαστε στα πλαίσια της διακυβέρνησης ε, των ε, οικονομικών περιόδων και θέλουμε να εντάξουμε τη συνθήκη αυτή σε ένα κοινοτικό πλαίσιο λαμβάνοντας κυρίως υπόψη την ευελιξία η οποία είναι τμήμα του πακέτου σταθερότητας. στόχος είναι να ενισχύσουμε πάντα τον δημοκρατικό έλεγχο και εδώ φυσικά ο έλεγχος θα μπορεί να γίνεται και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με το Fiscal Board, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Είναι σαφές ότι θα αξιολογεί τον τρόπο εφαρμογής των κανόνων που διέπουν ε, ε, τα δημοσιονομικά θέματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο αλλάζει τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον έλεγχο ας πούμε της δημοσιονομικής πολιτικής των κρατών μελών. Και εγώ να προσθέσω λίγα στοιχεία εδώ Αυτά θα αρχίσουμε να τα συζητάμε στην ουσία από το Δεκέμβριο, αλλά για την απλοποίηση φυσικά δεν θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τότε η συζήτηση. Θα πρέπει να συζητήσουμε και μετά τις συναντήσεις για το 2 και το 6-pack στις αρχές του επόμενου χρόνου. Είναι σαφές ότι δεν υπάρχει μία μόνο μορφή απάντησης η οποία να μας δώσει αυτόματα λύσεις και γι' αυτό ακριβώς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώνουμε τα όρια τα οποία έχουμε αλλά πρέπει τον ρόλο μας να τον ολοκληρώσουμε αν θέλετε και νομίζω ακριβώς γι' αυτό το λόγο ότι οι δυνατότητες που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην εποπτεία των προϋπολογισμών θα πρέπει να διατηρηθούν πλήρως. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριος Γκουαλτιέρη. Θα πρέπει να τελειώσουμε εδώ. Ο κύριος Καλβέτ Σαμπον για ένα λεπτό. Γρήγορα παρακαλώ γιατί κλείνουμε. Να υπενθυμίσω, λέει ο κύριος Καλβέτ Σόμπον, ότι δεν είναι σωστό να λέγεται ότι ε, η Ισπανία δεν καταθέτει προϋπολογισμό διότι υπάρχει θέμα με την Καταλωνία κτλ. Αν θέλετε πράγματι να προσφέρετε υπηρεσίες στον Ισπανικό λαό, να μην δεχθείτε παρακαλώ αυτή την ανακατανομή, την ανόητη των ευθυνών που προσπαθεί να κάνει η Ισπανική κυβέρνηση. Αυτό δεν είναι κάτι το ξαφνικό. Η κατάσταση σήμερα προετοιμάζεται εδώ και δεκαετίες. Υπάρχουν λοιπόν δύο θέματα σε επίπεδο δημοσιονομικό το οποίο πρέπει να απαιτήσετε πρώτον η εφαρμογή σωστή της ενιαίας αγοράς και δεύτερον μια ριζική ανακατανομή ε, των πόρων σε περιφερειακό επίπεδο. Νομίζω ότι δεν λειτουργείται ε, σε καιρούς οι οποίοι είναι ε, υπερβολικά φιλελεύθεροι. Κοιτάξτε, δεν ισχύει κάτι τέτοιο όπως είπατε, λέει ο κύριος Μοσκόβηση. Εγώ δεν είμαι εδώ για να κρίνω την πολιτική κατάσταση στην Καταλωνία, την κατάσταση που ισχύει σήμερα, το προηγούμενό της και τις συνέπειές της. Απλά προσπαθούμε να εξηγήσουμε ότι στην παρούσα φάση δεν υπάρχει δυνατότητα κατάθεσης ενός πλήρους προϋπολογισμού και γι' αυτό κάναμε την διάκριση ανάμεσα στον ισπανικό προϋπολογισμό ε, και στην Αυστρία και τη Γερμανία όπου τα πράγματα είναι διαφορετικά. Όλοι όμως έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι θα κατατεθεί η πρόταση σε ένα μικροχρονικό διάστημα και από τη Γερμανία και την Αυστρία το ταχύτερο δυνατόν σεβόμενοι πλήρως τους κοινοτικούς κανόνες. Σας ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος, θα κλείσουμε εδώ. Πράγματι οι αρμοδιότητες της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι σαφέστατες στη συγκεκριμένη περίπτωση. Διαπιστώνουμε τα όρια τα οποία υπάρχουν. Βλέπουμε και κάποιες πιθανές αντιφάσεις που μπορεί να υπάρχουν με τη συνθήκη και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί. Σας ε, ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας εδώ. Τέλος.